Okay, could you take your seats, please? Καλό καθίστε, καθίστε αν θέλετε. If you, if take your seat. Αν θέλετε, καθίστε. Και τις κάρτες σας να τις βάλετε τώρα στο μηχάνημα. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ελπίζω ότι όλοι έχετε τις κάρτες σας. Βλέπω πόσοι ψηφίζουν προτού προχωρήσουμε για να έχουμε το σωστό αριθμό που θα συμμετέχουν. Ανοίγεται η συσκευή. Λοιπόν, άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Αν θέλετε ψηφίστε όλοι σας. Όλοι είναι Εντάξει, ψηφίσατε όλοι εκτός μικροφώνου. Otherwise, say that we. It, it, it, it wasn't a real vote, so it doesn't matter. Another one? No, no, no, no. But when we come to the first vote, when it says plus one over on the it tells you, yeah. It showed plus one. Yeah, yeah it showed plus yeah, one. You could warn that already. Right. Okay. I just like to warn. Εντάξει. Θέλω να σας προειδοποιήσω ότι είναι μια ομάδα που έχει έναν παραπάνω από αυτούς που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Όταν θα περάσουμε στην πραγματική πλέον ψηφοφορία θα του το πω να αφαιρεθεί αυτός. Πρώτα απ' όλα, έγκριση ημερήσιας διάταξης. Ούντο, παρακαλώ. Πρόεδρε, αυτά που έχουμε σήμερα στον κατάλογο είναι πολλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη. Και είναι η πρώτη έκθεση οικονομικής στρατηγικής πολιτικής όπου το Ευρωκοινοβούλιο έχει διαδικασία συναπόφασης, συναποφασίζει από πλευρά του. Για την ομάδα μου θα ήθελα να πω ότι σε όλους τους εισηγητές και όλους τους κοιόδης εισηγητές εκφράζουμε ευχαριστίες που πολλές ώρες δουλειά επένδυσαν. Όμως δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτό το σημείο όπου αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μπορούμε να ψηφίζουμε ενιαία ενωμένοι. Κρίμα. Δεν θα έχουμε μεγάλες πλειοψηφίες για μια στρατηγική τοποθέτηση από πλευράς μας, που είναι όμως σημαντική υπόθεση στην αντιπαράθεση στις διαβουλεύσεις πραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ όμως για την κινητοποίηση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες και ευχαριστώ τους συναδέφου που συμμετείχαν σε αυτές τις προσπάθειες και ιδιαίτερα όσον αφορά την συνάδελφο Βότμαν Κορ. Ανταποκριθήκαμε ένα στον άλλο κινηθήκαμε ένα προς τον άλλο. Αλλά εκείνοι που ήθελαν να περάσουμε πέρα από την κρίση, να την ξεπεράσουμε και το σύμφωνο σταθερότητας να γίνει σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξη, εκείνοι που επιθυμούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική του 2020 να είναι πιο δεσμευτικοί αυτοί οι στόχοι από ό,τι μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάποιο συμβιβασμό σχετικά και γι' αυτό θα ήταν ε, νομίζω αξιόλογο, θα άξιζε να είχαμε λίγο χρόνο να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το συμβιβασμό. Προτείνω να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία λοιπόν πρόεδρε, ώστε να μπορέσει αυτό το Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει με μια ενιαία, ενωμένη φωνή όταν θα έχουμε την εκπροσώπηση των συμφερόντων της Ευρώπης την επόμενη εβδομάδα στις διαπραγματεύσεις. Θα ήταν πραγματικά κρίμα αν ψηφίζαμε απόψε και αποδυναμώναμε έτσι το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Jean-Paul, Jean εσείς ζητησατε τον λόγο παρακαλώ. Jean-Paul Ευχαριστώ. Άκουσα την πρόταση του κύριου Μπούλμαν, πρέπει να πω. Και θα ήθελα να πω ότι η δική μου ομάδα είναι υπέρ να ψηφίσουμε σήμερα. Να το εξηγήσω γιατί είμαστε υπέρ του να ψηφίσουμε σήμερα. Διότι το Συμβούλιο σε αυτό το χαρτοφυλάκιο εργάστηκε εδώ και πολύ χρονικό διάστημα και βρήκε λύσεις από πλευράς του. Τώρα, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε το δυνατόν πιο σύντομα να τοποθετηθεί από αυτών των προτάσεων για να καταλάβουν οι πολίτες μας περί τίνος πρόκειται και ποιον ρόλο διαδραματίζουμε εδώ. Τώρα, αν η αναζήτηση συμβιβασμών ήταν κάτι το οποίο θα επεκτηνόταν στο διηναικές, Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να οδηγήσει να επιτευχθούν όμως παρόλα αυτά κάποιοι τέτοιοι συμβιβασμοί σύντομα, δεν θα, πετυ... δεν θα βελτιώναμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια τη θέση του το Ευρωκοινοβουλίο εναντί του Συμβουλίου, ώστε να αναζητηθούν δυνατότητες για το μέλλον η τοποθέτησή μας για την οικονομία, η οικονομία μας να ενισχυθεί και τα αναγκαία μέσα να χρησιμοποιηθούν, ώστε οι οικονομίε μας και η ανάπτυξη να έχουν καλύτερα θεμέλια. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλο θα ήθελε να λάβει τον λόγο για αυτό το θέμα. Τότε, δεδομένων των συνθήκων, θα το θέσω σε ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρότασή μου είναι να συνεχίσουμε, να ψηφίσουμε δηλαδή, να συνεχιστεί η διαδικασία. Να αρχίσει λοιπόν η ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα για το αν επιθυμούμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του Ούντο Μπούλμαν να αναβληθεί. Αν ψηφίσετε ναι, υπέρ λοιπόν της αναβολής, αν ψηφίσετε κατά, τότε θα σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία επ' αυτού. Right, we've got one... Α, εντάξει, έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ και έναν παραπάνω από την, ε, τους σοσιαλιστές. Είναι δυνατόν να διευθετηθεί αυτό. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορία, λοιπόν. Και απορρίφθηκε η πρόταση. Λοιπόν θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. 17 υπέρ, 28 εναντίον. Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε λοιπόν. Έχω μια ανακοίνωση της Πρόεδρου. Δηλαδή θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση του κανονισμού για τι διασυνοριακέ μεταφορές μετρητών σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη έκθεση Και σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι οι διαπραγματεύσει στέφθηκαν με επιτυχία και ολοκληρώθηκαν με τη γραπτή διαδικασία και οδήγησαν σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Η Κορεπέρ θα υιοθετήσει το κείμενο της πρότασης στις 4 Μαΐου. Εκτός αν υπάρξουν ενστάσεις από την ομάδα αυτήν στον συμβιβασμό, τότε το σχέδιο Έκθεση θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιουνίου, στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου. Δεν υπάρχουν λοιπόν υποθέτω ενστάσεις. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η ανάγνωση και αυτή η συμφωνία στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου. Περνάμε τώρα το πραγματικό ψητό της συνάντησής μας, <laughs> της συνεδρίασής μας για απόψε. Λοιπόν, εντάξει. Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, Ούντο, εσείς πάλι παρακαλώ, χωρίς μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα για την ψηφοφορία. Θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, γιατί ουσιαστικά εκπροσωπούμαστε με τέτοιους αριθμούς ε, μελών όπως απαιτείται. Θέλω να αποφύγω κάποιες αμφιβολίες. Πριν ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία, να γίνει δοκιμαστική ψηφοφορία, να καταμετρήσουμε τα μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν από πλευρά των κοινοβουλευτικών ομάδων στον αριθμό τους. Να το ελέγξουμε. Πρόεδρος, Ευχαριστώ να κάνω και άλλη μια ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Αλλά κάθε μία έδειχνε ότι υπήρχε ένας παραπάνω. Ένας παραπάνω και ανεφάθηκε και από ποιους. Θα σας πω αν κάποιος ε, παρισφρήσει και χρησιμοποιήσει την κάρτα του ψηφίζοντας χωρίς να έχει δικαίωμα. Ας το κάνουμε όμως, δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε για να δούμε τον αριθμό. 50 κάρτες έχουμε, δύο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. 48 θα έπρεπε να ήταν το σύνολο. Right. EP. Λοιπόν, το ΕΛΚ έχει δύο παραπάνω μέλη, εντάξει. Το ΕΛΚ έχει δύο παραπάνω ακόμα. Δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα. Τώρα εντάξει, τώρα έχουμε 48 που συμμετέχουν με τις κάρτες τους. 47, 48 τώρα κάρτες. Τρεις δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία καθόλου, γιατί δεν έχουν πατήσει τα κουμπάκια τους. Υποθέτω εσκεμένα, έτσι. We've got three cards Τρεις έχουν βάλει τις κάρτες τους αλλά δεν συμμετέχουν πατώντας το κουμπί στην ψηφοφορία. It doesn't matter because they're not surplus to requirements. It's just... Είναι απλώς ότι κάποιοι δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, λίγη αυτή η ψηφοφορία εν πάση περιπτώσει. Και τώρα θα σας πω τι κάνουμε. Θα ψηφίσουμε με τη σειρά των εκθέσεων όπως συζητήθηκαν σε κάθε μία από τις συνεδριάσεις μας. Με τη σειρά λοιπόν της ε, ε, εκθέσεις Κόλ ε, ε, και στη συνέχεια Φεϊό, Φερέρα και τα λοιπά. Η Βόρτμαν Κόλ τώρα πρώτα θα ψηφίσουμε την έκθεση της Βότμαν Βόρτμαν Κόλ. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε την ψηφοφορία για το αν θέλουμε να απορρίψουμε το σύνολο ή όχι. Και μετά θα ψηφίσουμε για την νομική βάση ξεχωριστά και μετά από αυτές τις ψηφοφορίες θα περάσουμε στις λεπτομέρειες για την πολιτική, θέματα που έχει εξετάσει ήδη η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, η πρόταση απόρριψης, η τροπολογία για απόρριψη 66 και 67 που είναι ταυτόσιμες θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία. Οι οι σοσιαλιστές έχουν έναν παραπάνω ξαφνικά πάλι τώρα. Πρέπει να, να απορριφθεί η ψηφοφορία και να ξαναρχίσουμε. Έχουμε έναν παραπάνω πάλι. Ξαναρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Right, Okay, okay. vote's Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε. 42 εναντίον, 4 υπέρ. Και τώρα θα περάσουμε στη νομική βάση. Τροπολογία 68 και 69, 1 και 69, άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκαν. 18 υπέρ, 28 εναντίον. Και έτσι θα περάσουμε και θα ψηφίσουμε την τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 40 εναντίον, 6 υπέρ. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό Α. Έχουμε σε τμήματα ψηφοφορία. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Από το this μέχρι το του employment. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 45 υπέρ. Ένας εναντίον. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 28 υπέρ 18 εναντίον. Περνάμε στον συμβιβασμό Β. Όλο σε ένα τμήμα. Όλοι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία διορθώνει πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 46 υπέρ. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό γάμα C. Έχουμε προφορική τροποποίηση εδώ από τους σοσιαλιστές να αντικατασταθεί το procedural διαδικαστικά από το institutional διαθεσμικά. Γίνεται δεκτό, δεκτό. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 41 υπέρ και 5 εναντίον εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό ΔΔ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 19 εναντίον εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ και 16 εναντίον. Περνάμε στο συμβιβασμό ε σε ένα τμήμα ολόκληρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 27 υπέρ 19 εναντίον εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στον συμβιβασμό σίγμα F σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 30 in 16 υπέρ 16 εναντίον. Εγκρίθηκε. Well, that's, that's, that's a bit of excitement. We've opened Το θα πει αγωνία. Άρχισε η ψηφοφορία λοιπόν για το πρώτο τμήμα και εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα τώρα του συμβιβασμού σίγμα ταφ F. Άρχεται η ψηφοφορία δεύτερο τμήμα του F του σίγμα ταφ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αυτό εγκρίθηκε. 30 υπέρ 16 εναντίον. Περνάμε στον συμβιβασμό ZG. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 45 υπέρ 1 εναντίον εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 30 υπέρ 16 εναντίον. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό ΙΤΑ H σε δύο τμήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 16 εναντίον. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο ακόμα να ψηφίσουν. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Έληξη ψηφοφορία. 29 υπέρ 16 εναντίον. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό Ιώτα. Σε δύο τμήματα. Άρχεται στο πρώτο τμήμα πρώτα. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 7 εναντίον Άρχεται η ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα. Λίγη, σε λίγο η ψηφοφορία. Έληξε 27 υπέρ 19 εναντίον εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό J. Σε ένα τμήμα ολόκληρο άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 28 υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό και συμβιβασμός και σε ένα τμήμα ολόκληρος άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 28 υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στο R παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το R. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 2 εναντίον. M, συμβιβασμός σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 3 ε, εναντίον εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ 16 εναντίον. Συμβιβασμός 1, Στη συνέχεια δύο τμήματα Άρχεται η ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. 33 υπέρ 3 εναντίον. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ υπέρ και 15 εναντίον εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό O, ΙΣΤΑΦ 16. Σε ένα τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ 7 εναντίον. Περνάμε στο συμβιβασμό τον 17 άρχεται η ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Ε, όλο ένα τμήμα με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 15 εναντίον. Πάμε στην τροπολογία 383. Φαίνεται είναι δική μου αυτή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Δεν είσαστε αρκετά θαραλέοι. Αυτό είναι το πρόβλημα φαίνεται. Καταψηφίστηκε. Θα το μετανιώσετε. Συμβιβασμός Q. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 36 υπέρ 5 εναντίον πέντε αποχές. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. 27 υπέρ το αποτάσμα 12 εναντίον 7 αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στον συμβιβασμό Α. Ιωτα θήτα. Σε ένα τμήμα ψηφίζουμε Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφόρειας. 30 υπέρ 14 εναντίον. Δύο αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 438. Άρχεται η ψηφοφορία για την 438. 438. 438 Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 16 υπέρ, 28 εναντίον, μία αποχή. Τα καταφέρατε καλύτερα από μένα, Φιλίπ. 439 τροπολογία τώρα. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 8 εναντίον μία αποχή. Βίκη, συγχαρητήρια, τα πήγατε καλά. Συμβιβασμός σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Συμβιβασμός λάμδα S. Το πρώτο τμήμα ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. 41 υπέρ, 4 εναντίον εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα του S του λάμδα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 26 υπέρ, 19 εναντίον. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό λάμδα α. Τι ψηφίζουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ 18 εναντίον μία αποχή Πάμε τώρα στον συμβιβασμό U22 λάμδα β. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ 19 εναντίον. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό v 23 σε ένα τμήμα, λάμδα Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 44 υπέρ 2 εναντίον. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό W24. Άρχεται η ψηφοφορία λάμδα δέλτα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ 15 εναντίον. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό 6. Άρχεται να το βρω πρώτα και άρχεται η ψηφοφορία τώρα λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, 41 υπέρ, 3 εναντίον, 2 αποχές. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό Y. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, 27 υπέρ 19 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό Z. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 29 υπέρ 14 εναντίον 3 αποχές. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό AA, σε ένα τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 42 υπέρ 2 εναντίον 2 αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 549, 549. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 31 υπέρ 14 εναντίον εγκρίθηκε. Καλύτερα τα πάω τώρα εν πάση περιπτώσει. Συμβιβασμός, μια στιγμή. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ομού τις επόμενες τροπολογίες 952, 52, 53 από κοινού θα ψηφίσουμε 550, 551, 552, 553 αυτές τις τέσσερις τροπολογίες. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα να ψηφίσουν. Μια στιγμή. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Τέλος. Και αποτέλεσμα τέσσερις υπέρ 42 εναντίον. Απορρίφθηκαν. Τώρα περνάμε στον συμβιβασμό ΑΒ σε ένα τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ ένας εναντίον, δύο αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβασμό AC, ΑΓ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τελευταία ευκαιρία για σας τους δύο. 41 λοιπόν, 41 υπέρ, μία, ένας εναντίον, δύο αποχές. Περνάμε στον συμβασμό. Όχι, όχι. Πάμε στην τροπολογία 555. 555 πρώτα. Άρχεται. Ένας ακόμα έβαλε την κάρτα του και ψηφίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 18 υπέρ 28 εναντίον απορρίφθηκε Λυπούμε Σιλβί, δεν τα κατάφερες. Συμβιβασμός ΑΔΕΛΤΑ, AD, ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα, 43 υπέρ. Ένας εναντίον, δύο αποχές. Το δεύτερο τμήμα τώρα της ΑΔΕΛΤΑ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τελευταία ευκαιρία. Τέλος ψηφοφορία τώρα. Αποτέλεσμα 31 υπέρ, 3 εναντίον. 3 εναντίον, 12 αποχές. Και περνάμε στην τροπολογία 558. Τροπολογία 558. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε αυτή με 14 ψήφους υπέρ 32 εναντίον. Καμία αποχή. Ε, περνάμε τώρα στην 559 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε και αυτή 16 υπέρ 28 εναντίον Δύο αποχές. οι τροπολογίες 71, 72, 73 είναι ταυτόσιμε για τις αιτιολογικέ σκέψεις, τις ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 27 υπέρ 17 εναντίον. Δύο αποχές εγκρίθηκαν. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό ΑΕΕ. Ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Mm. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 30 υπέρ 14 εναντίον 2 αποχές. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό α ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 29 υπέρ, 17 εναντίον, άλλαξε. 30 είναι υπέρ και 16 εναντίον. Πατήσατε το λάθος κουμπί για την ΑΣΤΑΦ, την ΑΕΦ, γι' αυτό. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον συμβιβασμό αζ-AG. Σε ένα τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 3 εναντίον εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό AH, α, ή άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. 43 υπέρ, ένας εναντίον, δύο αποχές. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό AI, άρχεται η ψηφοφορία. αλφα αλφα-ιτα ψηφίσατε όλοι Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 15 εναντίον και Περνάμε τώρα στο AJ. Α, δηλαδή. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 13 εναντίον, 2 αποχές. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 28 υπέρ 17 εναντίον μία αποχή. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό AK. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ 18 εναντίον μία αποχή. Περνάμε στο συμβιβασμό AR στη συνέχεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελευταία ευκαιρία να ψηφίσετε και τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 41 υπέρ, 2 εναντίον, 2 αποχές. Εγκρίθηκε, περνάμε στο συμβιβασμό AM και ψηφίζουμε, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 31 υπέρ, 15 εναντίον εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό AN. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 13 εναντίον, 2 αποχές εγκρίθηκε. Τώρα Έχουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε που πρέπει να ψηφίσουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 27 υπέρ, 18 εναντίον, μία αποχή. Και τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 27 υπέρ, 18 εναντίον, μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Βότμαν Ζητήσατε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έδωσαν μια δυνατή πλειοψηφία σε μένα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε μια πρόταση όπου θέλουμε να έχουμε και ισχυρή νομισματική και ισχυρή οικονομική ένωση. Κρίμα που οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για μια βιώσιμη ε, δημοσιονομική εποπτεία. Όλοι οι συγκητές έχουν τη λεξούλα τους. Προχωρούμε. Έκθεση Φέιο. Καθίστε καταρχάς, έξι εκθέσεις έχουμε. Όπως και πριν, μπαίνουμε πρώτα στα διαδικαστικά. Τροπολογίες 51-52. Για απόρριψη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 4 υπέρ 41 κατά. Νομική βάση τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 52. Ψηφίσατε, Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 3 υπέρ 43 κατά. Χειρότερο από απόρριψη κύριε Αντιπρόεδρε. Η πλατφόρμα δεν έχει καλή αντιμετώπιση σήμερα. Συμβιβαστική Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 2 κατά. Προχωρούμε. 165 το υπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Προχωρούμε. 24 τροπολογία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ 12 κατά μία αποχή. Καταπίπτουν οι υπόλοιπες τροπολογίες μέχρι την 26. 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρα στις ψηφοφορίες. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Τροπολογία 169 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ε, ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. 4 υπέρ 41 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Άρα τροπολογία 170. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία, 15 υπέρ 30 κατά μία αποχή. Και αυτή η τοπολογία απορρίπτεται. 171. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ 16 κατά δύο αποχές. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική Β τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Προχωρούμε στην 187. 187 τροπολογία. ψηφίσετε όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 16 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική γάμα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 3 κατά. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 18 κατά. Προχωρούμε. 201 τροπολογία, ενώ υπάρχει και μια προφορική τροπολογία του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ 15 κατά 3 αποχές. 202 και 203 τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται, Πέρας. 14 υπέρ 31 κατά 1 αποχή. Απορρίπτεται. 204 ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. 205. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ 31 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. 206. ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ 13 κατά 2 αποχές. 207 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική Δέλτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. 25 υπέρ 17 κατά 4 εποχές. 212 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ 16 κατά, οι δύο εποχές. Συμβιβαστική ε. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 42 υπέρ 3 κατά και μία εποχή. Δεκτή. Συμβιβαστική σίγμα ταφ. F. Ψηφίσατε όλοι υπέρ της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 17 κατά δύο αποχές. ...225 τροπολογία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφι υπέρ, 13 κατά μία εποχή. 31.1 πρώτο τμήμα και 224 που είναι όμοιες. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 2 αποχές. 227 Λάθος το έκανα. Ψηφίζουμε 327. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. «29 υπέρ 15 κατά 2 αποχές». Είπα ότι είναι ίδιες. Όχι σωστό, σωστό. Όχι, δεν έκανε τίποτα λάθος. 228. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορία. 44 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Δεκτή. 229 Πέρα Πέρας ψηφοφορία. 43 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. 32 το υπολογία. Ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική Ζ, G, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 39 υπέρ 5 κατά 2 αποχές. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία, 29 υπέρ 15 κατά 2 αποχές. Συμβιβαστική ΙΤΑ H με μια προφορική τροπολογία. με προφορική τροπολογία του κ. Σικλούνα. Θέλετε να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Άρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία μόνο. 17 υπέρ 26 κατά δύο αποχές για την προφορική τροπολογία. Τώρα η συμβαστική λύση χωρίς την προφορική τροπολογία, το συμβαστικό κείμενο. Ένας ΕΛΚ παραπάνω είναι. Ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ 6 κατά για το βασικό κείμενο συμβιβασμού H, ήτα. ΆΙ, τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορία. 44 υπέρ. 1 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική πρόταση J, J, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 42 υπέρ 3 κατά. Δεύτερο τμήμα. Ψήφισετε όλοι πέρα της 28 28-18. 225. Υπέρ, ψηφίζουμε. Ψήφισετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 41 υπέρ 2 ε, κατά 2 εποχές. Καταπίπτει 37. Συμβιβαστική ΚΑΠΑ, ΙΑ. κέι δηλαδή, ΙΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 16 κατά. 38 τροπολογία. Ψηφίσετε όλοι. 43 υπέρ, κανένας κατά δύο αποχές. Γυρίζουμε σελίδα. Συμβιβαστική L, ΙΒ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ μία αποχή. Συμβιβαστική M ΙΓ με προφορική τροπολογία του κύριου Σικλούνα. Τη δεχόμαστε? Ψηφίζουμε χωριστά τη συμβιβαστική τοπολογία; Την προφορική τροπολογία, συγγνώμη. Αυτό κάνουμε αν δεν γίνεται δεκτή μια προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε μόνο την προφορική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 26 κατά δύο εποχές για την προφορική τοπολογία. Άρα δεν θα συμπεριληφθεί στο συμβιβαστικό κείμενο. Ψηφίζουμε τώρα την συμβιβαστική τροπολογία MJΓ. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 38 είπε ρεπτάκατα. Συμβιβαστική πρόταση N, δέλτα Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συμβιβαστική O, ΙΕ Άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 39 υπέρ 6 κατά. Καμία αποχή. Συμβιβαστική π. Ιώτα σίγμα Ψηφίζουμε την συμβιβαστική π λατινικό Ιώτα σίγμα ελληνικό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Τροπολογία 272 και 273 που είναι ίδιες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ 30 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία του εισηγητού 45. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε κι άλλες κι άλλες ψηφοφορίες. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ 17 και δύο αποχές η τροπολογία 17 της Επιτροπής Απασχόλησης. Συμβατή λέει. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 26 κατά, δύο εποχές. Συμβιβαστική Q, λατινικά γιοταζίτα. Ψηφίζουμε την πρόταση αυτή. Ψηφίσατε όλοι υπέρ τη ψηφοφορία, 44 υπέρ, μία κατά, μία αποχέ. 276 τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, 43 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Δεκτή. 277 και 278 τροπολογίες ίδιες ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας 14 υπέρ 31 κατά μία αποχή απορρίπτεται η 19 της Επιτροπής Απασχόλησης ψηφίζουμε Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ, καμία κατά, δύο αποχές. 20, ε, συγγνώμη, 279 τροπολογία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 2 υπέρ, 43 κατά, μία αποχή. 20 της Επιτροπής Απασχόλησης, ψηφίσατε όλοι, Πέρα της ψηφοφορίας, 43 υπέρ, μία κατά, δύο αποχές, συμβιβαστική R, γιώτα τα ελληνικά, ψηφίσατε όλοι, Πέρας το 32 υπέρ 12 κατά. ...283 και 284 τροπολογίες που είναι ίδιες, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ 31 κατά μία αποχή. 285 ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας 17 υπέρ 28 κατά μία αποχή απορρίπτεται συμβιβαστική S φύτα ελληνικά ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας. 44 υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Συμβιβαστική ταφτί λατινικά κάπα, κοστί ελληνικά. Διορθώνει πρόεδρος, πρόκειται για μία ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα της συμβαστικής αυτής προτάσεως, ψηφίζετε όλοι, πέρας ψηφοφορία. 42 υπέρ τρεις κατά. Το δεύτερο τμήμα, η φράση, Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 15 κατά. Καμία αποχή. 292. Τροπολογία. Ψηφίζεται. Πέρας. 14 υπέρ 31 κατά μία αποχή απορρίπτεται. 293. Ψηφίζεται όλοι, πέρα ψηφοφορία. 17 υπέρ, 28 κατά μία αποχή. 294. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δύο υπέρ 43 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται 300 το υπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Κανείς δεν είναι υπέρ. 43 κατά 3 εποχές. Μα ο κόσμος ψηφίζει κατά των τροπολογιών που καταθέτει. Ωραίο αυτό. 295. Ψηφίζεται όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 2 υπέρ. 43 κατά μία αποχή. 296 τροπολογία. Ψηφίσετε, πέρας πληροφορίας. 15 υπέρ, 30 κατά μία αποχή. Κατοπίπτη. 298. Ψηφίσετε, πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, Επτά κατά, μία αποχή, δεκτή. Άρα η 299 διοθόνη, η 297 καταπίπτει, η 299 συμβατή και την ψηφίζουμε τώρα. 299 το υπολογία. Ψηφίσετε. Πέραση της 17 υπέρ 28 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική U, ΚΑ στα ελληνικά, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 42 υπέρ 4 κατά. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσετε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 38 υπέρ 8 κατά καμία εποχή. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε την 50. Everybody's voted, 44 υπέρ, δύο αποχές, κανείς κατά. Η, 210, η 310 συγγνώμη είναι συμβατή. Ψηφίζουμε την 310 υπολογία. Votes closing, votes closed. 42 in favor. 42 υπέρ, 2 κατά μία αποχή. Δεκτή. Συμβιβαστική πρόταση Β λατινικό, ΚΒ ελληνικό. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβαστική W, ΚΓ ελληνικά, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 27 κατά 2 αποχές. Καταπίπτει. Τροπολογία 63. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ μία ψήφος κατά μία αποχή. Δεκτή. 64. Has everybody voted? Votes Ψηφίσατε όλοι. 41 ψήφοι υπέρ, 2 ε, κατά και μία αποχή δεκτή. 65 αποσύρθηκε, 68. Ψηφίσατε όλοι. 42 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. 69 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίες. 27 υπέρ 14 κατά 4 αποχές. Τώρα προχωρούμε στη συμβιβαστική XKΔ ελληνικά. ψηφισετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 72-1-1 Πέρας ψηφοφορίας 42, 1, 1. Εβδομήντα τέσσερα. Πέρας ψηφοφορίας. Δύο υπέρ 43 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. 75. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 7 υπέρ 38 κατά καμία εποχή. 76. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Τρεις υπέρ 39 κατά τρεις αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Y, Ε. ελληνικά. Ψηφίζετε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφι υπέρ, 15 κατά καμία αποχή. Τροπολογία 3, Ψηφίζεται όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ 16 κατά μία αποχή. Καταπίπτει η 85. Συμβαστική Z. Κάπα σίγμα τάφ. όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. 87 άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 87 πέρας ψηφοφορίας 40 υπέρ 5 κατά μία αποχή ευχαριστώ συμβιβαστική AA καπαζίτα 42-2 δεκτή. Συμβιβαστική πρόταση ΑΒ ΚΙ ελληνικά. closed. 45 in favor. 45 υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 υπέρ, 14 κατά, 2 αποχές. Αλφασί συμβιβαστική και άλλη οριζόντια συμβιβαστική ψήφισαν όλοι. Πατήστε το κουμπάκι, πέρας. 42 υπέρ, 3 κατά, χωρίς αποχές τροπολογία 8. Ψήφισαν όλοι πέρας. 45 υπέρ, κανείς κατά και μία αποχή. Η 102 καταπίπτει, πάμε στη συμβιβαστική ΑΔ, ε, Ψήφισαν όλοι, πέρας. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική ΑΕ ΕΙ. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική AF, ε, ΑΕ Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, 14 κατά μία αποχή. Τώρα, 105 τροπολογία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 43 υπέρ, 1 κατά μία αποχή. 106. Α, 106 μέχρι 110 όλες μαζί. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί, 106 με 110. Και Εκα... Α, δεν θέλουν. 106. Υπέρ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 40 υπέρ 4 κατά μία αποχή. 107 Α, τώρα μπορούμε να κάνουμε όλες μαζί, 107 με 110, όλες μαζί τις ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 35 υπέρ, 9 κατά και μία αποχή για όλες αυτές, μέχρι και την 110. 111. Ψήφισαν όλοι πέρας. 3 υπέρ 42 κατά μία αποχή. Τον 11 πέρας. 28 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Είναι 112 αυτό. 100 την AG συμβιβαστική τώρα. Ψήφισαν όλοι πέρας. 43 υπέρ, 2 κατά, χωρίς αποχές. 113 τροπολογία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. 114. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 14. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 15. Ψήφισαν όλοι πέρας. 43 υπέρ, 3 κατά, χωρίς αποχές. Συμβιβαστική AH. Ψήφισαν όλοι πέρας. 45 υπέρ, κανείς κατά, κανείς αποχές. Αλλά δύο δεν πάντησα, πάντησα το κουμπάκι η συμβαστική AI. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 44 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. 124. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Συμβιβαστική AJ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 42 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. 22 υπέρ, 23 κατά και μία αποχή καταπίπτει. Αυτό ήταν το πιο μικρό αποτέλεσμα, 134 ψήφισαν όλοι πέρας. 26 υπέρ 19 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική AK. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 38 υπέρ 6 κατά 2 αποχές. 138 Ψήφισαν όλοι. Ψηφίζουν κι άλλοι. 43 υπέρ. Ένας κατά. Μία αποχή. Την την 139 δεν θα την ψηφίσουμε γιατί έχει γιατί ψηφίστηκε η 134. Πάμε στην 140. Ψήφισαν όλοι την 140. Πέρας. 39 υπέρ. 2 κατά. 5 αποχές. Πάμε στην 142. Ψηφίζουμε την 142. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Πε, όχι, τώρα πέρας. 42 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. 143. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 39 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. 144. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 33 υπέρ, 13 κατά, χωρίς αποχές. Πάμε στη συμβιβαστική AL. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Πάμε στη συμβιβαστική AM τώρα. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. 46 υπέρ χωρίς ψήφους κατά ούτε αποχές. 150. Ψήφισαν όλοι πέρας. 14 υπέρ 31 κατά με μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν και πάμε στην 151 τροπολογία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 44 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. 152. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 3 υπέρ, 42 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. 153. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 υπέρ 3 κακά 2 αποχές. 154 καταπίπτει. Πάμε στην 20. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ 13 κατά μία αποχή. Οπότε καταπίπτουν οι υπόλοιπες και πάμε στην τροπολογία 158. Το ΕΛΚ έχει μία παραπάνω. Ξέρω ότι είναι η Άστριντ αλλά ξέρω κάποιος πρέπει να, να κάνει πίσω. Έτσι, μείον μία. Εντάξει τώρα. 42 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εντάξει. Κάποιος μένει πιστός. 21, τροπολογία 21. Η τροπολογία 21 από τον εισηγητή ε, πέρας 42 υπέρ 3 κατά μία αποχή τροπολογία 22 πέρας 44 υπέρ 1 κατά μία αποχή οπότε πάμε τώρα στην 23 Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 38 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Τώρα θα πάμε... Καταπίπτει 159, πάμε στην συμβιβαστική αλφανή σε δύο τμήματα. Η πρώτη είναι η πρώτο, πρώτο τμήμα της ΑΕΝ. Ψήφισαν όλοι. Παρακαλώ. Πέρας. Τελειώνουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 38 υπέρ και 4 κατά. Δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 37 υπέρ 8 κατά χωρίς αποχές. Λοιπόν, ψηφίζουμε το κείμενο όσο τροποποιήθη. Ένας ψήφος, μια ψήφος ΕΛΚ περισσεύει. Ε, κάποιος συμμετέχει ενώ δεν πρέπει. Ευχαριστώ. Οπότε είμαστε 29 υπέρ, 7 κατά και 10 αποχές. Και ψηφίζουμε τώρα και το νομοθετικό ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι πέρας. 28 υπέρ 7 κατά και 11 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κύριος Φέιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Θα είμαι σύντομο. Δεν είναι τώρα χρόνος για μεγάλες πολιτικές δηλώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα μέλη του γραφείου μου, τους βοηθούς μου, για την προσπάθεια που κατέβαλαν να γίνει καλά αυτή η δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική μου ομάδα, το ΕΛΚΑ και την Κορίν Βότμαν Κόλ που και η γραμματεία είχαν κύριο ρόλο. Σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές ευχαριστίες που είχα ευκαιρία μαζί τους με διαφορετικές αφετηρίες να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους. Τους υπόλοιπους εισηγητές ευχαριστώ πολύ για αυτό το πακέτο εκθέσεων. Οι συναντήσεις μας θα συνεχιστούν ελπίζω και σύμφωνα με την αρχή αυτή όπως πάντα που ακολουθούμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Προεδρείο, την Πρόεδρο και τη Γραμματεία για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Και θέλω να ολοκληρώσω με δύο λόγια όσον αφορά εκείνους που πάντα είχαν ε, τοποθέτηση κατά ή καταψήφισαν για αυτή την έκθεση και όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν στην Ολομέλεια θα προσπαθήσω να τους πείσω και να τους πείσω να υπερψηφίσουν και όχι να καταψηφίσουν. Και με αυτή την ελπίδα θέλω να ευχαριστήσω όλους και πάλι θερμά. Um, Ευχαριστώ πολύ. Σιλβίκο, ξέρουμε και βλέπουμε ότι παίρνουν χρόνο οι ψηφοφορίες. Μη διαβάζετε ίσως τα αποτελέσματα, να εξοικονομήσουμε λίγο, να λέμε μόνο ε, δεκτό ή απορρίπτεται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Μην διαβάζουμε τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε δύο πίνακες που τα βλέπουμε εμείς από εδώ. Και εγώ ήθελα να πω, παρόλο που ζούμε σε περίοδο λιτότητας, να παπιούμε λίγο καφέ να μας προσφερθεί. Θα γίνει μετά την τρίτη ψηφοφορία ένα μικρό διάλειμμα. Τώρα θα κάνουμε την τρίτη ψηφοφορία. Δεν χάνω χρόνο γιατί πρέπει να τα καταγράψουμε τα αποτελέσματα και πρέπει να ξαναρχίσει να, να τεθεί σε λειτουργία πάλι το μηχάνημα για τις ψηφοφορίες, την ηλεκτρονική ψηφοφορία, οπότε δεν χάνουμε χρόνο θέλω να σας πω που τα διαβάζουμε. Είπαμε από την αρχή ότι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τα πάντα, αυτό δεν αλλάζει, δεν το αλλάζω εγώ. Τώρα θα πάμε στην έκθεση Φερέιρα, όπου θα αρχίσουμε με την απόρριψη της πρότασης άρχεται η ψηφοφορία. απόρριψη δηλαδή τη πρόταση της Κομισιόν. Ψήφισαν όλοι. Παρακαλώ, η ψυχά μας δυσκολεύεται γιατί τα ακούμε όλα έτσι όπως είναι η κατασκευασμένη αίθουσα. Κάποια μέλη λείπουν. Δεν συμμετείχαν. Τέλο πάντων, ε, τελειώνουμε πέρα τη ψηφοφορία. 3 υπέρ, 41 κατά, χωρίς αποχές. Τώρα προχωρούμε. Νομική βάση που είναι συμβιβαστική, είναι συμβιβαστική α, α, μείον α, συμβιβαστική μείον α λέγεται. Η συμβιβαστική μείον α λοιπόν ψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Προχωρούμε τώρα Μισό λεπτό. Στην 50. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 50. Ψήφισαν όλοι πέρας. 3 υπέρ, 40 κατά και μια αποχή. Πάμε στην τροπολογία 1 ε, από την Επιτροπή ε, Προσχώρησης. Ψήφισαν όλοι πέρας. 18 υπέρ 23 κατά και 2 αποχές. Συμβιβαστική Α. Γρήγορα με τα κουμπάκια. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Κλείνουμε όμως. 43 υπέρ 1 κατά. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική Β. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής τροπολογίας Β. Παρακαλώ μην ε, κάνετε φασαρία. Ψήφισαν όλοι. Τελειώνουμε πέρα της ψηφοφορίας. 40 υπέρ 3 κατά αποχές. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική Σ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε τη συμβιβαστική ΣΥ. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 42 υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Και πάμε τώρα στην 190. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 24 υπέρ 19 κατά. Πάμε στη συμβαστική δέλτα, D. Ψήφισαν όλοι. Τελειώνουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 42 υπέρ 1 κατά. Η 203 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 203. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 16 υπέρ 27 κατά. Απορρίφθηκε με μία αποχή. Συμβιβαστική ε ή. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 41 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Και πάμε τώρα στην 223. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 223. Μάλιστα. 2-2-3. 2-2-3. Δεν είναι αυτό στην, ε, στον κατάλογο του εισηγητή που έχω εγώ. Αυτό που λέτε εσείς δεν είναι στο δικό μου κατάλογο. Ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε. Τελειώνει η ψηφοφορία. Απερίφθη τέλο πάντων 20 υπέρ 22 κατά 225. Ψηφίσατε πέρας. 40 υπέρ 4 κατά μία αποχή συμβιβαστική F ε, ψήφισαν όλοι πέρας 44 υπέρ χωρίς αποχές και ψήφους κατά πάμε στη συμβιβαστική G άρχεται η ψηφοφορία G. Πέρας. 39 υπέρ 6 κατά. Τώρα πάμε στην επόμενη συμβιβαστική H σε 7 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το πρώτο της συμβιβαστικής H. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 υπέρ, 5 κατά. Δεύτερο τμήμα. Εψήφισαν όλοι πέρας. 40 υπέρ, 5 κατά. Τρίτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι πέρας. 22 υπέρ 22 κατά, αυτό καταπίπτει. Απορρίπτεται θέλω να πω. Πάμε στο τέταρτο τμήμα. Ε, ψήφισαν όλοι πέρας. 40 υπέρ 5 κατά. Πάμε τώρα στο πέμπτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι, πέρας. 39 υπέρ 5 κατά. Έκτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι, πέρας. 39 υπέρ 5 κατά μία αποχή και το έβδομο τμήμα Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 υπέρ και 5 κατά. Τώρα θα πάμε στην συμβιβαστική ΆΗ. Συμβιβαστική ΆΗ. Ζαν Πολ, τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν ε,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 Je suis là. I've got an amendment 247. You got that? 247. It seems to have disappeared. Ψάχνουμε την τροπολογία 247 και δεν τη βρίσκουμε.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 It's still there. It's there, but it's too late. Yeah. It's now included within yeah. the Madame, Madame la Présidente, pour, yeah. pour les membres du PPE. Εξ ονόματος των μελών του ΕΛΚ θα ήθελα να πω κάτι, δύο λόγια. Στρέφομαι στα μέλη του ΕΛΚ για να τους πω κάτι. Ο κατάλογος που έχουμε εδώ για την ψηφοφορία. Είναι παλαιότερος κατάλογος. Έχουμε έναν άλλον που ετοιμάστηκε κατά το απόγευμα. Ε, για κοιτάξτε, Ντόρφμαν έχει το ενισχύ κείμενο ο κύριος Ντόρφμαν και επ' αυτού θα μπορεί να γίνεται αναφορά. <laughs> yeah. Right. The, the, the problem was we Καλά, το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε χάσει μια τροπολογία που μετακινήθηκε όμως και τη βρήκαμε. Ήταν μια τη Σίλβια. Πριν από την ε, συμβιβαστική τώρα θα την ψηφίσουμε. Ξέχασα που είμαστε. Πού είμαστε. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική I, Ι, ακόμα μπορούμε να ψηφί... μπορείτε να ψηφίσετε. Αν δεν έχετε ψηφίσει την... επί της ε, συμβιβαστικής Ι, τελειώνετε παρακαλώ. Ωραία. Τώρα, πέρας της ψηφοφορίας 42 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. 2.45. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 21 υπέρ 22 εναντίον χάθηκε λοιπόν καταψηφίστηκε μία αποχή. Και πάμε στην τροπολογία 248. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 6 υπέρ 37 εναντίον μία αποχή. Καταψηφίστηκε συμβιβασμός J. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 41 υπέρ 2 αποχές. Πάμε λοιπόν στον συμβιβασμό και στη συνεχεια Α, ΙΑ11 στα ελληνικά. Ψηφίσατε όλοι. Συνεχίστε, πιέστε τα κουμπάκια όταν, όσο προλαβαίνετε. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Ψήφισαν 43 υπέρ ένας εναντίον. Περνάμε στο L. 12. ΙΒ. Συμβιβασμό L. Ψηφίσατε όλοι. Τέρμα ψηφοφορίας. 42 υπέρ. Κανείς εναντίον μία αποχή. Περνάμε στον συμβιβασμό M. 13 ΙΓ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 44 υπέρ, ένας εναντίον, ε, μια εποχή. Περνάμε στο συμβιβασμό N, 14 Ι δέλτα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ, ένας εναντίον. Καμία αποχή εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβίβα. Συντροπολογία 23 πρώτα. 23 Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέρμα ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 36 υπέρ. Κανείς εναντίον μία αποχή. Περνάμε στον συμβιβασμο ο ΙΕΟ15. Άρχεται. Ο15 ΙΕ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 42 υπέρ 1 εναντίον 2 αποχές. Περνάμε στην τροπολογία 269. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 17 υπέρ 26 εναντίον. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός π 16 ταφ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ, ένας εναντίον, μία αποχή. Και περνάμε στον συμβιβασμό Q17, ΙΖ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όλοι λέω. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ, 2 εναντίον, καμία αποχή. Περνάμε στον συμβιβασμό R, ΙΙ, 18 ψη... Φύσατε όλοι. Όλοι λέω. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 40 υπέρ 4 εναντίον μία αποχή. Περνάμε στην τροπολογία 284. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 21 υπέρ 22 εναντίον κατά ψηφίστηκε μία αποχή. Συμβιβασμός τώρα S στη συνέχεια 19 Ι.Θ. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 44 υπέρ. Μία αποχή εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 285. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 42 εναντίον καταψηφίστηκε πάμε στον συμβιβασμό T20 κάπα ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 43 υπέρ 2 εναντίον εγκρίθηκε και πάμε τώρα στον συμβιβασμό U21 καπα τι είναι αυτό εκεί Α, εντάξει η τροπολογία 247 σε σχέση με τον συμβιβασμό. Τι περνάμε στον γιου τώρα, συμβιβασμό γιου 21 κα Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 45 υπέρ, μία αποχή εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 290. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 20 24 εναντίον μία αποχή. Καταψηφίστηκε συμβιβασμός τώρα παρακαλώ 22 ΚΒ Β ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 44 υπέρ 1 εναντίον πάμε στον συμβιβασμό W ΚΓ 23 Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 44 υπέρ 1 εναντίον. Πάμε στον συμβιβασμό 624 ΚΔ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 41 υπέρ 4 εναντίον. Εγκρίθηκε και πάμε στο συμβιβασμό Y25 ΚΕ. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ 3 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στις ε, Επιτροπής Απασχόλησης 38. Employment 38. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 34, 34 υπέρ 9 εναντίον 2 αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 308. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Ε, τέλος ψηφοφορίας. 5 υπέρ, 37 εναντίον. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Z26 ε, ΤΑΦ Ψηφίσατε όλοι. Ελάτε, ξέρω ότι ήρθε καφές και αυτό σας ενδιαφέρει, αλλά παρόλα αυτά τα, τα κουμπάκια να πατάτε. Θα ολοκληρωθεί τώρα η ψηφοφορία επί του 26, τροπολογίας 26, αποτέλεσμα 44 υπέρ, ένας εναντίον. Περνάμε στον συμβασμό ΑΑ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της ΑΑ άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ 1 εναντίον. Δεύτερο τμήμα της ΑΑ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 22 υπέρ 22 εναντίον. Ισοψηφία καταψηφίστηκε. Χωρίς μικρόφωνο. Οι διερμηνείς δεν το άκουσαν. Εντάξει, θα ξαναψηφίσουμε. Ε, εδώ υπήρξε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το αντίτυπο. Ξεκινάμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Τώρα ψηφίζουν 46 από εσά. Εντάξει, λίγη ψηφοφορία. Διαβάστε τι είναι το δεύτερο τμήμα. Μπορείτε. Μόλις το ψηφίσαμε και καταψηφίστηκε 23 υπέρ τώρα και 24 εναντίον σε αυτή την ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα που ζητήσατε. Θέλετε να ακούσετε πραγματικά τι καλύπτει, πώς έχει διατύπωση. Πρόεδρε, μπορείτε, μπορούμε να επαναλάβουμε γιατί πραγματικά είχε δημιουργηθεί μπέρδεμα να το ξαναψηφίσουμε. Τι ψηφίζαμε το δεύτερο τμήμα ουσιαστικά η τελευταία ψηφοφορία ήταν για το δεύτερο τμήμα, το ξαναψηφίσαμε δεύτερη φορά και δύο φορές καταψηφίστηκε. Ισοψηφία η πρώτη 22-22, 23 υπέρ 24 εναντίον στη δεύτερη ψηφοφορία, πάλι καταψηφίστηκε. Απλά και μόνο επεξήγησα τι συνέβη. Αν πιστεύετε ότι υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, όπως είπατε, καθώς είχα και αυτό το πρόβλημα εγώ ως εισηγήτρια, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να επαναλάβω την ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα, για τη συμβαστική τροπολογία ΑΑ. Άρχεται τώρα και πάλι η ψηφοφορία για την ΑΑ τροπολογία. Εντάξει τώρα λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας. Και τώρα και πάλι 23 υπέρ 24 εναντίον. Αυτή τη φορά τρεις φορές καταψηφίστηκε αυτό. Ελπίζω να το αποδεχτείτε τώρα και με την τρίτη καταψήφιση. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 324 και 300. Ελίζα Φερέιρα, ησυχία παρακαλώ οι άλλοι. 46 ή 47, γιατί αυτό ήταν η ερώτηση μου. 48 είμαστε, αλλά ποτέ δεν ήταν 48 όλοι. Είχαμε μεταξύ 44 και 46 σε σχέση με τις ψηφοφορίες που συμμετείχαν. Εγώ περίμενα πάντα για να δω πόσοι θα πατούσαν το κουμπάκι, άφηνα πάντα επαρκή χρόνο να ψηφίσουν όλοι. Κάποιοι οι οποίοι όμως δεν ψηφίζουν, αλλιώς θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, 324 τροπολογία. Τώρα έχουμε 49 που ψηφίζουν. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ όμως. Λοιπόν, εντάξει. 48 τώρα κάρτες. 45 έχετε ψηφίσει ήδη. Έχουμε τώρα 46. Ένας παραπάνω όμως από το ΕΛΚ. Ένας από το ΕΛΚ πρέπει να αφαιρεθεί, να φύγει από όσους συμμετέχουν. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πάλι Τώρα εντάξει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορία τώρα. 17 υπέρ, 27 εναντίον. Καταψηφίστηκε η τροπολογία 324. Πράγμα που τώρα μας κάνει να πάμε στην 326. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 17 υπέρ 27 εναντίον μία αποχή καταψηφίστηκε. Συμβιβασμός Α2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 38 υπέρ 7 εναντίον μία αποχή εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα του ΑΒ συμβιβασμού άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας τώρα έληξε η ψηφοφορία αποτέλεσμα 39 υπέρ 5 εναντίον 2 αποχές Πάμε τώρα στον συμβιβασμό ΑΓΑΜΑ-AC σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα του ΑΓ συμβιβασμού άρχεται. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Θα σταματήσω μόνο όταν θα ησυχάσετε. Εντάξει, τώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 39 υπέρ 7 εναντίον. Δεύτερο τμήμα τώρα του ΑΓ συμβιβασμού. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Τελειώνει η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 36 υπέρ 6 εναντίον εγκρίθηκε. ΑΔ συμβιβασμός. AD άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 44 υπέρ, ένας εναντίον μια αποχή εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 339. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 38 υπέρ 6 εναντίον. Μία αποχή εγκρίθηκε. 340 τώρα τροπολογία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 17 υπέρ 26 εναντίον. Δύο αποχές. Καταψηφίστηκε. Συμβιβασμός ΑΕ. Ε, άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 44 υπέρ, ένας εναντίον μια αποχή. Πάμε στον συμβιβασμό AF, ΑΣ τάφα. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ όμως πάλι. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την ΑΣ συμβιβαστική τροπολογία, AF. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ, ένας εναντίον εγκρίθηκε. AG τώρα ο επόμενος συμβιβασμός, ΑΖ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ. 3 <clears throat> αποχές εγκρίθηκε. Ε, H, α ή τα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 45 υπέρ, μία αποχή εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία της ΑΙΤΑ συμβιβαστική. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 4 εναντίον. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό AI, ΑΘ. Άρχεται η ψηφοφορία για την ΑΘ, AI. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορία. 42 υπέρ, 2 αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην συμβαστική AJ, ΑΙ, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 39 υπέρ, 4 εναντίον, 3 αποχές. Δεύτερο τμήμα της ΑΙ, AJ, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ 5 εναντίον μία αποχή εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην AK συμβιβαστική τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Ελάτε, έχουμε άλλες 7 και ολοκληρώνουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 40 υπέρ 3 εναντίον 2 απόχέ εγκρίθηκε. Πάμε στην AL συμβιβαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. τέλο ψηφοφορία. 43 υπέρ 2 εναντίον 1 αποχή εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 39. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το Έλκο. Μόλις έβαλε την κάρτα του και πάτησε την τελευταία στιγμή το κουμπάκι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία και πάλι. 39 τροπολογία. Συνεχίζουμε επαναλαμβάνοντας την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 26 υπέρ, 17 εναντίον. Και πάμε στην τροπολογία AM. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 44 υπέρ, ένας εναντίον, μία αποχή, εγκρίθηκε. Πάμε στην AN τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 39 υπέρ 6 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 388. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 5 υπέρ 39 εναντίον. Απορρίφθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό AO. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ 3 αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό AP. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 43 υπέρ 3 αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 391 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Κλείνει η ψηφοφορία. Ελάτε. 17 υπέρ 25 εναντίον. Καταψηφίστηκε τροπολογία 392. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Ελάτε. Πέντε δεν έχουν ψηφίσει. Λίγη τώρα σε λίγο η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 16 υπέρ 26 εναντίον καταψηφίστηκε. 395 τροπολογία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 21 υπέρ 24 εναντίον καταψηφίστηκε. 396 τροπολογία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 22 υπέρ 23 εναντίον. Καταψηφίστηκε. 393 και 43. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία Και αποτέλεσμα 18 υπέρ 27 εναντίον καταψηφίστηκαν. Τροπολογία 394. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορία, 26 υπέρ 19 εναντίον εγκρίθηκε. Τροπολογία συμβιβαστική AQ. AQ μάλιστα. Συμβιβαστική IQ. Είναι στην επόμενη σελίδα μετά στον κατάλογο. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τελευταία ευκαιρία. Τώρα λίγη ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 43 υπέρ 1 εναντίον. Εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό AR. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 28 υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό AS. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 45 υπέρ. Μία αποχή εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στον συμβιβασμό AT. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 46 υπέρ. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός AU. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 46 υπέρ και εγκρίθηκε. Συμβιβασμός AW. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 45 υπέρ. Μία αποχή εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 407 μια στιγμή. Καταπίπτει λέει αν έχει εγκριθεί η προηγούμενη. Ωραία. Μάλιστα. Η 407 κατέπεσε λοιπόν σαν συνέπεια τούτου. Συμφωνεί ο εισηγητή. Περνάμε στον συμβιβασμό AX. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. τέλο ψηφοφορία Αποτέλεσμα 43 υπέρ εγκρίθηκε και ένα εναντίον. Δεύτερο τμήμα τώρα της AX. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 22 υπέρ 23 εναντίον μία αποχή καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε. Πάμε στην τροφολογία 410. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία τώρα. Έληξε η ψηφοφορία τελικά. Αποτέλεσμα 41 υπέρ, 3 εναντίον, εγκρίθηκε. Πάμε στο συμβιβασμό AY, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 43 υπέρ, 3 εναντίον, εγκρίθηκε και πάμε στην τροπολογία 61. Ψηφίσατε όλοι. τέλο ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 39 υπέρ. 5 εναντίον. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 58 και 4 τροπολογία Επιτροπής Απασχόλησης άρχονται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 35 υπέρ 10 εναντίον εγκρίθηκαν της απασχόλησης 5, employment 5. Ψηφίσατε όλοι. 17 υπέρ 27 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 60 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 41 υπέρ. 1 εναντίον. Εγκρίθηκε. Της απασχόλησης 6. Employment 6 αυτή κατέπεσε, λέει, εφόσον έχει η προηγούμενη εγκριθεί. Τροπολογία 59, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 34 υπέρ 10 εναντίον εγκρίθηκε. Της απασχόλησης η τροπολογία 3, employment 3. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ 11 εναντίον εγκρίθηκε. Συμβιβασμός AZ άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 43 υπέρ 2 εναντίον εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 68. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 5 εναντίον. Εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό BA. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 25 υπέρ, 20 εναντίον. Εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 25 εναντίον. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Πάμε τώρα στην τροπολογία 69. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 69, τροπολογία 69. Παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. 41 υπέρ 3 εναντίον. Τροπολογία 70. Άρχεται. Ομού να τις πάρουμε. Να τις πάρουμε από την 70 μέχρι την 74 όλες μαζί. 70. Ε, μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού εκτός από την 74. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε πιο γρήγορα αν τις πάρουμε με τη σειρά. 70 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 41 υπέρ 4 εναντίον εγκρίθηκε 71. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 44 υπέρ εγκρίθηκε 72. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 40 υπέρ και 4 εναντίον εγκρίθηκε. 73 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. 21-21 ισοψηφία απορρίφθηκε. Τροπολογία 74 τώρα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Ελάτε παρακαλώ. Σβέλτα, τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 17 εναντίον. Εγκρίθηκε. Η ΒΒ Συμβασική τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζεται πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 3 κατά. Δεύτερο τμήμα. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. 39 υπέρ 6 κατά. Το υπουργείο 78. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 7 κατά, 17 ε, κατά. 79 Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ 21 κατά. Τροπολογία 80. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. Η 9 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας ψηφοφορίας. 34 υπέρ 9 κατά. Τροπολογία 81. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 82. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ 14 κατά. 83 Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 15 κατά. 84 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. 85 Ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 8 κατά, δεκτή. 86. Πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 3 κατά. 87 Ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 22 κατά. Απορρίπτεται. 88. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 23 κατά αποτρίπτεται 89. Πέρας ψηφοφορίας. 9 υπέρ 35 κατά. 90. Δεν έχουμε χρόνο. Εάν δεν πάμε πιο γρήγορα θα χάσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται. 10 επιτροπή Απασχόλησης. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ 5 κατά. 91. Κάντε κάτι για να πιέσετε λίγο πιο γρήγορα τα κουτιά, τα, τα κουμπιά σας, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 15 κατά. 92 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. 8 ε, κατά, δεκτή 93. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ. 17 κατά, 11 ε, ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορία. 17 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται. 12 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 27 απορρίπτεται. 94 Ψήφισαν όλοι πέρας. 39 κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική BC σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. 37 προς 8. Εντάξει δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίφθηκε αυτό. Τρίτο τμήμα. Τελειώνουμε την ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό αυτό. Τέταρτο τμήμα τώρα. Το τέταρτο τμήμα ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη αυτό. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική BD σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απερίφθη αυτό. 22 προς 25, τρίτο τμήμα. Ησυχία παρακαλώ. Τελειώνουμε πέρας. Δεκτό αυτό. Τέταρτο τμήμα. Άλλοι ψηφίζουν. Τελειώνουμε. Δεκτό αυτό. Πέμπτο τμήμα. Πέρας. Απερίφθη το αυτό, 22 προς 25. Πάμε στη συμβιβαστική BE. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτή, 41, προς... πάμε στο 106. Απερίφθη αυτό. 107 Πέρας. Δεκτό, 23 προς 21. Ησυχία, παρακαλώ. Αν θέλουμε να τελειώσουμε τις ψηφοφορίες σήμερα, πρέπει να τελειώνουμε. BF, συμβιβαστική BF, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό 43 προς 3. Δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη 14 προς 32. Και το τρίτο τμήμα. Πέρας. 41 προς 5 δεκτό. Πάμε τώρα στην 113 τροπολογία. Και ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 114. Εψήφισαν όλοι. Περισσεύει ε, μία ψήφος ΕΛΚ. Πέρας. Εντάξει. Απερίφθη. Συμβιβαστική BG. Τελειώνουμε. Πέρας. 42 υπέρ 3 αποχές. Πάμε στην 122. Ψήφισαν όλοι, τελειώνουμε, πέρας, δεκτή, 39 προς 5, η 6 τώρα, που είναι, 123, ψηφίζουμε την 123. Εψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή 40 προς 4. Η 18, γνωμοδότηση ΕΜΠΛ, δεν ψηφίζουμε τη 18. Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 18 προς 25. 124. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή 39 προς 5. 125. Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 17 προς 28 έχει καταπέσει 6. Πάμε στην 126. Η 126. Εψήφισαν όλοι. τελειώνουμε. Τώρα περισσεύει μία ψήφος ΕΛΚ. Ποιος έχει ψηφίσει. Ωραία. Ευχαριστώ απερίφθη αυτή 18 προς 27 ή 127. Τελειώνουμε πέρας. Απερίφθη 16 προς 28. Τροπολογία 19 από την απασχόληση. Α, έχει καταπέσει αυτή. Ε, όχι. Δεν έχει καταπέσει. 19 ε, της απασχόλησης. Εδώ είμαστε. Πέρας. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Τώρα έχει καταρριφθεί, απορριφθεί. Προχωρούμε στην τροπολογία 7. Καταπίπτει αν κάτι έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει εγκριθεί μάλλον. <laughs> Πέρας. Απερίφθη αυτή, 22 προς 23, η 128 τώρα τίθεται σε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 23 προς 23. Η 129 Περισσεύει πάλι μια ψήφος ΕΛΚ. Mm, πολύς ενθουσιασμός βλέπω, αλλά ας βγει κάποιος από το ΕΛΚ παρακαλώ. Εντάξει, πέρας. Αυτή απορρίφθηκε 21 προς 22. Η, η τροπολογία 130 τώρα. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Αυτή εγκρίθηκε 27 προς 17. Τώρα, η τροπολογία 131. Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 17 προς 28. 132. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Απερίφθηκε αυτή η 17 προς 27, τροπολογία 8. Εψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή 40 προς 5. Η 134 ψηφίζουμε. Εψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 31 προς 2 135 Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Δεκτή 27 προς 18. Συμβιβαστική BH. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε δεκτή 40 προς 5. Πάμε τώρα στην 139. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Απερίφθη 17 προς 27. 140. Εψήφισαν όλοι πέρας απερίφθη 19 προς 26, 141. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. 17 προς 28. Πάμε στην Employment 20, από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Εψήφισαν όλοι. Πέρας απερίφθη 16 προς 28 142 Εψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή. 37 προς 7. 143. Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 17 προς 28, 145. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Πέρας. Απερίφθη 15 προς 28. Η 9 έχει καταπέσει. Πάμε στην 144. Ψηφίζουμε. Την 144 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή 42 προς 1. Η 146 κατέπεσε. 147 ψηφίζεται. Τίθεται σε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή 29 προς 16. 148. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 37 προς 9. Δεκτή. Συμβιβαστική BI. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 43 προς 2. Πάμε τώρα στην 153 τροπολογία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθει αυτή, 20 προς 24. Η 154. Περισσεύει μια ψήφος ΕΛΚΑ. Συνεχίζετε να αποπειράστε. Πέρας. 25 προς 17 δεκτή. 155 Εψήφισαν όλοι πέρας. Αυτή απερίφθη 21 προς 23. 156. Πέρας. Απερίφθη 19 προς 27. Ε, employment 22. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 15 προς 28. 157. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 17 προς 28. Employment 23. Ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή. 39 προς 6. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν έτσι, ε. Μέχρι την 160. Αυτή θα την ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίζουμε την 160. Εψήφισαν όλοι. Συνεχίστε. Εντάξει, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας. Απερίφθη αυτή. 10 προς 21 ψήφους. 161. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 43 προς 1. 163. Εψήφισαν όλοι. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπάκια. Παρακαλώ, ελάτε, ακόμα 7 έχουμε, πέρας, δεκτή 29 προς 13, 164. ψήφισαν όλοι. Πέρας. 43 προς 1 δεκτή. Τώρα, επόμενη είναι η 167. Ψηφίζουμε επί της 167 τροπολογίας. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 27 προς 18. Employment 24. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη 17 προς 26. Συμβιβαστική BJ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Εψήφισαν όλοι πέρας δεκτό 43 προς 3 και το δεύτερο τμήμα εψήφισαν όλοι πέρας δεκτό 41 προς 5 τώρα το, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε δεν φτάσαμε ακόμα εκεί ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε τώρα περισσεύει μια ψήφος ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πέρας. 42 υπέρ 4, 4 κατά αποχές δεκτό λοιπόν. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Συνεχίστε να ψηφίζετε, δεν έχουμε όλες τις ψήφους. Εντάξει, τελειώνουμε πέρας της ψηφοφορίας. 41 προς 4. Κάποιον χάσαμε στο ενδιάμεσο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να δούμε και το χρόνο, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ελίζα. Θα δώσω το λόγο σύντομα πολύ στην Ελίζα. Ξέρω ότι όλοι έχουμε κουραστεί πια. Ζητώ όμως συγγνώμη. Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω επανειλημμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθερή πλειοψηφία για να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Αυτό χάρη στη δουλειά των σκιωδών εισηγητών και ιδιαίτερα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον Καρλ Άγκλοντ που έχει την έκθεση που ακόμα θα ψηφίσουμε και που είναι εταίρος αυτή η έκθεση της δικής μου έκθεσης. <laughs> οι άλλοι εισηγητές που εργαστήκαμε από κοινού νομίζω με αποτελέσματα που μπορούν ακόμα να βελτιωθούν περαιτέρω και τη γραμματεία ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία της δικής μου κοινοβουλευτικής ομάδας ή της γενικής, τη Γενική Γραμματεία της ε, Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της δικής μου κοινοβουλευτικής ομάδας διότι έκαναν πολλές προσαρμογές ε, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν την ε, ιδιότητά μου ως εισηγήτρια στην έκθεσή μου αυτή. Ευχαριστώ. Right, colleagues, we are going to... Ωραία. Συναδελφοί, θα φύγουν οι διερμηνείς. Προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε, ξέρετε όλοι τι γίνεται, ακόμα θα έχουμε τους διαρμηνείς. Προχωρούμε στην έκθεση Γκουλάρ, όπως πριν. Παρακαλώ. Είμαστε τώρα στην έκθεση Γκουλάρ 55, 56, 57 που απορρίπτουν το, την πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη λοιπόν. Δεν θα ψηφίσουμε την 96. Πάμε στη νομική βάση. Ε, τροπολογέν. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή 35 προς 8. Τροπολογία 58. Ψήφισαν όλοι. Συνεχίστε να ψηφίζετε. 10 δεν έχουμε ακόμη ψηφίσει. Τελειώνουμε την ψηφοφορία. Την κλείνουμε καταπίπτει 19 προς 19. Και πολλοί δεν ψηφίσατε. Οι 180. Unblock. όλες μαζί. Μέχρι την 186. 180 προς 186 όλες μαζί. somebody can't. which one can't you? Μισό λεπτό. Τι μπορούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτές τις έξι τροπολογίες. Πέρας. Ποια? Τις πρώτες τρεις. Μαζί. Μπορείτε. Άρα τις πρώτες τρεις, με 180 με 182. just you know it, we waste more time trying to deal with the blocks. Okay, now we've got one too many EPP. Έχουμε έναν ELK παραπάνω. Κάποιος από το ELK. Right. The vote's closed. Right, that's rejected by 40 to 3. Right, we now... 3 υπέρ 40 κατά απορρίπτεται. Το 184 μόνο του. Το Τροπολογία 184 μόνη τη. Μέχρι την 186. 184 186. Μαζί. Voted. Five if you haven't. I'm closing the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 προς 29. 187. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3 υπέρ 41 κατά. Συμβιβαστική α σε δύο τμήματα. Ψηφίσετε. Τέλος ψηφοφορίας για το πρώτο. Δεκτό. 41 προς 4. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσετε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 41 προς 5 επίσης. 199 τροπολογία και 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 2 υπέρ, 43 κατά. 35. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 36 προς 3, καταπίπτουν οι λοιπές. 207 τώρα. Ψήφισατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 12 προς 30. Συμβιβαστική Β. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 38 προς 6. 220. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 προς 26. Συμβιβαστική γάμα. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή, 44 προς 1. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 31 προς 1. Τρίτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 42 προς 3. 246 τροπολογία. Ψηφίζουμε για την 246. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3 προς 42. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 41 προς 3. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. 17. 27 προς 7. 263 τροπολογία. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3 προς 42. Συμβιβαστική ε σε 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. 43 δεκτή. 43 εδώ. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 28 προς 6. Τρίτο τμήμα. Περαιώνουμε την ψηφοφορία. Δεκτή 27 προς 6. Τέταρτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή 39 προς 6. Πέμπτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας δεκτό 27 προς 18. Τροπολογία 286. Κάποιος έλκα εξτρά θα κάθεται κάπου, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Εντάξει. Άλλοι πέντε πρέπει να ψηφίσουν. Ψηφίσετε. Απορρίπτεται. 15 προς 27. 287. Ψηφίσατε. Απορρίπτεται. 3 προς 42. 288. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται σε 14.31. 2.89. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 προς 30. 21 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 προς 28. Συμβιβαστική F. Σίγματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό το τμήμα το 36-3. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορία Δεκτό 36 προς 9. 2.97 το απολογία. Όχι, έχει καταπέσει. Ζήτα. G σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό 42, σε δεκτό τμήμα, 42 προς 1. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 43 προς 3. 53 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. 36 προς 1 δεκτό. Συμβιβαστική ήττα σε ένα τμήμα αλλά με μία προφορική τροπολογία. Θέλουμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την προφορική. Ψηφίζετε. Κάνα δυο. Ακόμα να ψηφίσουν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η προφορική τροπολογία. το συμβιβαστικό κείμενο αυτό καθεαυτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρες. Δεκτό το, δεκτή 27 προς 16. 298. το 298 και το 299 απορρίπτεται. Ε, συμβαστική θήτα I, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 40 προς 4 δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Όλο και πιο γρήγορα πάμε. Αλλά χρόνο θέλει ακόμα. Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορίε. Οκτώ δεν έχετε ψηφίσει ακόμα. Τέλο πάντων, δεκτό. 33 προ 5. Γιώτα, Τζέι. Πρώτο τμήμα. Δεκτό. 42 προς ένα Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. 23 προς 5. 13 αποχές. Συμβιβαστική Ι και δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, 37 προς 7. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 23 προς 20 δεκτό. Τρίτο τμήμα. Κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτό 38 προς 6. Τέταρτο τμήμα. Κλείνω. Δεκτό. 39 προς 6. Συμβιβαστική L, Α. δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας πληροφορίας. Δεκτό. 34 προς 7. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσετε. Κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτό. 35 προς 7. 307 τροπολογία. Ψηφίζετε, ψηφίζετε. Νωρίς και συχνά, λέμε εμείς στη Βρετανία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 προς 28 απορρίπτεται. Τροπολογία συμβιβαστική M, ΙΓ. Ψηφίζουμε. Κλείνω. Δεκτό. 40 προς 3. Τροπολογία 59. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 60. Ψηφίστε. Κλείνω. Κλείνω. Απορρίπτεται. 2 προς 43. 61. Κλείνω. Απορρίπτεται. 5 προς 38. 63. Περαιούται. Απορρίπτεται. 17 προς 28. Συμβιβαστική N, γιώτα Ψηφίσατε. Δεκτή. 42 προς 2. Συμβιβαστική όμικρον ο λατινικό, γιώτα ελληνικό. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 42 προς 2. Συμβιβαστική πι λατινική γιώτα σίγμα τάφ. Κλείνουμε. Δεκτή 42 προς 1. Συμβιβαστική Q. Γιώτα Ζ. Ψηφίσετε. Δεκτή 44 δύο εποχές. Τροπολογία 77. Ψηφίζουμε. Ψηφίζετε. Κλείνουμε. Απορρίπτεται. 15 προς 31. 78. Ψηφίζετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 37 προς 6. Καταπίπτει 8. 79. Ψηφίζουμε. Πέρας πληροφορίες απορρίπτεται. 17 προ 27. 80. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή. 37 προ 5. Συμβιβαστική R. Ιωταΐτα. Ψηφίσετε. Δεκτό το κείμενο 41 προς 4. Ένα της Επιτροπής Αποσχόλησης. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή 38 προς 5. Δύο της ίδιας Επιτροπής. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή. 35 προς 7. 84. Ψηφίσετε. Πέρας. Δεκτή. 43 με 2 αποχές. 85. Ψηφίσετε. Πέρας. Δεκτή 26 προς 18. Η 86 έχει αποσυρθεί. 88. Πέρας πληροφορίες για την 88 δεκτή. 29 προς 15. Συμβιβαστική S, γιώτα θήτα. Ψηφίσετε Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 40 προς 2. Συμβιβαστική τι. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 36 προς 7 δεκτή. Συμβιβαστική UKα. Ψηφίσατε. Πέρας πληροφορία. Δεκτή 40 προς 3. Συμβιβαστική Β, ΚΒ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή 40 προς 1. Τροπολογία 11. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 39 προς 2. Συμβιβαστική W Γ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέρμα. 42 υπέρ. Τροπολογία 97 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 98. Ψηφίσατε. Περαιούται. Απορρίπτεται. 8 προς 33. 99. Πέρας ψηφοφορία. 5 προς 38 απορρίπτεται. 12 Κλείνουμε, κλείσαμε. 34 προς 7, δεκτή. Άρα τώρα πάμε στην 102. Ψηφίσατε. Κλείσαμε. Απορρίπτεται. 14 προς 28. 3 της Επιτροπής Αποσχόλησης. Ψηφίζουμε την απασχόληση 3. Δεν πέρασε 102. Μισό, μισό. Λάθος, λάθος. Η 12 πέρασε. 103. Κλείνουμε. Δεκτή. 37 προς 6. 4 καταπίπτει. 104. Ψηφίσετε. Κλείσαμε. Απορρίπτεται. 6 προς 37. 5 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 προς 25. 105. Πέρας. Απορρίπτεται. 3 προς 40. 106. Πέρας. Δεκτή 35 προς 8. Καταπίπτει 13. Συμβιβαστική X δέλτα. Ψηφίσατε. Περαιούται. Περαιώθηκε. Δεκτή 33 προς 8. 108. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 προς 35. Y, ε, ε, κάπα, τι είναι αυτό τώρα, κάπα ε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Δεκτή τροπολογία 35 προς 8. Συμβαστική Z, κάπα σίγμα ταφ. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή 36 προς 6. 118 τροπολογία. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή 39 με καμία ψήφο κατά. Καταπίπτει 16. 120. Το Απολογία 120. Πέρας πληροφορίας. 36 υπέρ 4 κατά. 20 καταπίπτει. 124 για 125 ομού. Κλείνουμε, κλείσαμε. Απορρίπτονται 17 προς 25. 126. Ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίπτεται. 0 προς 40. 127. Ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 προς 23. 128. Ψηφίσετε. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. 2 προς 41. 129. Ψηφίσετε. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. 17 προς 24. 22 της εισηγήτριας. Ψηφίσετε. Κλείσαμε. Δεκτή. 31 προς 10. Καταπίπτουν οι 130 και 7. 131. 131. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή. 22 προς 16. 132. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 προς 27. 133. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή. 41 προς 3. 23 της ηγήτριας. Ψηφίσατε. Δεκτή. Συμβιβαστική αλφα-αλφα, δηλαδή ελληνικά ΚΖ. Ψηφίσατε. Πέρας. Δεκτή 41 προς 3. Η 135 τροπολογία. Ψηφίσατε. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. 136. Πέρας πληροφορίας δεκτή. 35 προς 6.

Δεν πάνε γρήγορα. Απορρίπτεται. 15 προς 29. 145. Πέρας. Απερίφθη 17 προς 26. 25. Ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 24 προς 19 9 146 καταπίπτουν πάμε στην 147 Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 3 προς 39. 148. Εψήφισαν όλοι πέρας. 39 προς 2. 149. Πέρας. Απερίφθη. 3 προς 40. Employment 10. Και ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη 8 προς 35 150 Εψήφισαν όλοι πέρας Απερίφθη 3 προς 41 154 Εψήφισαν όλοι πέρας Απερίφθη 5 προς 39

Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθησαν 8 προς 35. 160. Εκατόν εξήντα. Ένα έξι Κλείνουμε πέρας. Απερίφθη 17 προς 26. 161. Εψήφισαν όλοι πέρας. Απερίφθη 17 προς 26. 162. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 17 προς 27. 26. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 9 προς 35. Employment 11. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. 21 προς 21. 27. Ψήφισαν όλοι πέρας. Δεκτή 44 προς 1. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική Αλφαβήτα. δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο. Ψήφισαν όλοι πέρας. 37 προς 4 δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. 36 προς 9. Δεκτό και αυτό. Τώρα. 170. Εψήφισαν όλοι πέρας απορρίφθηκε 10 προς 34. 171. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίφθηκε 15 προς 30. Employment 13. Εψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 37 προς 5 172 ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 39 προς 6 173 Εψήφισαν όλοι πέρας, απερίφθη 3 προς 41. 174-175. Πέρας. Απερίφθησαν 15 προς 29. 176. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη 20 προς 23. Τροπολογία 29. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, κατα, απορρίπτεται 23 προς 23. 178. Πέρας. Καταπίπτει. Ε, απορρίπτεται. 3 προς 43. 177. ψήφισαν όλοι. Ελάτε. Πέρας. Απορρίπτεται 19 προς 24. 179. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 προς 26. Τροπολογία 30. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 30 προς 15. Τροπολογία 31. Ψήφισαν όλοι. Τελειώνουμε πέρας. Δεκτή 40 προς 1. Συμβιβαστική AC. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. τελειώνουμε. Πέρας. 42 προς 1. Δεκτή. Συμβαστική AD. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 41 προς 3. Συμβιβαστική ΑΕ. Πέρας. Δεκτή. 42 προς 4. AF ε συμβιβαστική. Λοιπόν, ένας παραπερισσεύει από το ΕΛΚ, να αφαιρεθεί παρακαλώ. Πέρας, δεκτή, 41, 41 ψήφι προς 2. Ψηφίζουμε τώρα επί του κειμένου ως έχει τροποποιηθεί. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουμε. Ένας, εντάξει ψηφίσατε όλοι, πέρασε. 33 υπέρ 14 κατά χωρίς αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Μία ακόμα ψήφος μας λείπει, εντάξει, πέρασε. 36 υπέρ 11 κατά χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια. Ωραία. Σάρον, μια λέξη πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ όλους. Συνεχίζουμε. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες ακόμη και όταν φύγουν οι διερμηνείς. Αλλιώς πρέπει να επανέλθουμε πρωί-πρωί πριν αρχίσει η επισήμωση Επιτροπή για να τελειώσουμε. Αύριο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για λόγους αρχής θέλω να εκφράσω μια ένσταση ότι μια ψηφοφορία, μια συνεδρίαση με ψηφοφορίες θα μπορεί να διεξαχθεί χωρίς διερμηνία. Αυτό είναι ένσταση δική μου. Αλλά τέλος πάντων, για σε σχέση με το που είπατε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και εγώ θλίβομαι γι' αυτό. Θα ευχόμουν να είχαμε περισσότερο χρόνο ώστε να μπορούσαμε να τα ολοκληρώσουμε. Αν κάποιος δεν τα καταφέρει θα έχει πρόβλημα. Ψηφίζουμε για την απόρριψη. Περνάμε τώρα στην έκθεση Hagland, δηλαδή με άλλα λόγια λέει η πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την απόρριψη, για την πρόταση απόρριψης. Όχι κατά την ψηφοφορία, δεν γίνεται τέτοια παρέμβαση. Πολύ φασαρία γίνεται παίρνει το λόγο ο μιλητή. Πρόεδρε, εξηγήστε μας τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε διερμηνία ή δεν θα έχουμε διερμηνία στη συνέχεια. Τι γίνεται. Δεν θα έχουμε διερμηνία είπατε μετά. Ε. Ε, γιατί δεν ψηφίζουμε αύριο τότε και συνεχίζουμε απόψε. Αύριο το πρωί μπορούμε, έχουμε συνεδρίαση, να συνεχίσουμε, να κάνουμε συνεδρίαση και να συνεχίσουμε. Ο συνάδελφος παρενέβη και το είπε, γιατί δεν μπορούμε αύριο να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Θα έχουμε διερμηνία και δεν θα υπάρχει πρόβλημα για κανέναν. Ουσιαστικά ρωτήσαμε, ο κύριος Γκοζέ. Διαμαρτύρομαι διότι δεν υπάρχει διερμηνία κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. Είπα ωστόσο ότι μπορούμε κατά εξαίρεση να συνεχίσουμε να ψηφίσουμε, ούτως ώστε όλοι οι παρόντες να μπορέσουν να μετάσχουν. Αύριο μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες να έχουμε επαρκή, επαρκή αριθμό μελών για την ψηφοφορία. Αυτή είναι η θέση μας. Λυπούμε λοιπόν, πρέπει να πω. Πιθανώς αυτή είναι η βούληση συντριπτικά των μελών και ρωτήσαμε πριν γίνει αυτή η αναγκαιρία. Θα το ψηφίσουμε αν επιθυμείτε, αλλά δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία θα ήθελε να συνεχίσουμε έτσι. Εσείς παρακαλώ. Ήδη έχουμε συζητήσει σε σχέση με τους ε, διερμηνείς, έχουμε ρωτήσει αν μπορούν να συνεχίσουν ή όχι. Και είπαν όχι, ε, θα συνεχίσουν. Θα ήθελα να ρωτήσετε λοιπόν, να συντάξετε μια επιστολή για αυτό το γεγονός δεσμεύονται από χρονικά όρια για τη δουλειά τους Γενικά είναι πολύ γενναιόδοροι, γενναιόδοροι οι διερμηνείς και δίνουν παράταση χρόνου όταν χρειάζεται. Όταν λήξει η διερμηνία, αν κάποιος έχει δυσκολία, ε, τότε θα το αναγγείλει και θα προσπαθήσουμε έτσι να το λύσουμε όπως θα γίνεται. Βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας ε, για την απόρριψη. Θα ψηφίσετε στο τέλος. Έξι από εσά δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Άλλοι που θα ψηφίσουν παρακαλώ θα λήξει τώρα η ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, απορρίφθηκε. 3 υπέρ 36 εναντίον. Απόρριψη λοιπόν. Περνάμε στην ε, νομική γνωμοδότηση. Ψηφίζουμε την νομική βάση για αυτό το θέμα. Τροπολογία 34. Νομική βάση 34. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 13 υπέρ, 26 εναντίον. Συμβιβασμός α, άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε 39 υπέρ, 3 εναντίον. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 159. 159 παρακαλώ. Άλλοι που θα ψηφίσετε τώρα για τη λίγη, έληξε λίγη ψηφοφορία, έληξε τώρα η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε λοιπόν 17 υπέρ 25 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 161. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε 15 υπέρ 25 εναντίον. Τροπολογία 162. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 41 εναντίον, 1 υπέρ. Τροπολογία 163. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 3 υπέρ, 37 εναντίον. Συμβιβασμός Β. Σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. 40 υπέρ, 3 εναντίον. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέσσερις ακόμα πρέπει να συμμετάσχουν για να ολοκληρώσουμε. Λίγη ψηφοφορία τώρα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε 38 υπέρ 2 εναντίον. Τρίτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέντε ακόμη πρέπει να ψηφίσουν και θα λήξει η ψηφοφορία. Έληξε 25 υπέρ 15 εναντίον. Τέταρτο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Θα λήξει τώρα η ψηφοφορία. Έληξε, εγκρίθηκε 37 υπέρ 5 εναντίον. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται. <clears throat> Τώρα θα λήξει η ψηφοφορία. Έληξε. Αποτέλεσμα 37 υπέρ 6 εναντίον. Εγκρίθηκε. Αυτό ήταν λοιπόν για το συμβιβαστικό Β. Έχουμε τώρα μια άλλη ψηφοφορία για το έκτο τμήμα το έκτο το οποίο αποκαλείται τμήμα 2 γιατί είχαμε σε το 2 να το ψηφίσουμε αυτό πρέπει έχουμε τα πέντε τμήματα το υπόλοιπο του κειμένου είναι το υπόλοιπο α εντάξει το υπόλοιπο του κειμένου να ψηφίσουμε λοιπόν έγινε υπόλοιπο κειμένου που δεν ψηφίστηκε σε τμήματα αυτό ψηφίζουμε λοιπόν το υπόλοιπο άρχεται το κατανοούμε τέλεια ψηφίσατε όλοι Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Συνεπές αυτό. Περνάμε στην τροπολογία 227 παρακαλώ. Σελίδα 8 στο δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας. Εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, τροπολογία 227 που ψηφίζουμε και άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απο... Καταψηφίστηκε 22 εναντίον 20 υπέρ. Αν είχα ψηφίσει, σωστά καταφέρναμε. Συμβασμός γάμα πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 36 υπέρ, 5 εναντίον. Δεύτερο τμήμα του γάμα, συμβιβασμού γάμα. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε 36 υπέρ 6 εναντίον. Συμβιβασμός Λι, παρακαλώ. Πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 38 υπέρ 3 εναντίον. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 41 υπέρ, 3 εναντίον. Πάμε τώρα στην τροπολογία 249. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 39 υπέρ, 4 εναντίον. Συμβιβασμός ε ή άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε 43 υπέρ 1 εναντίον συμβιβασμός F σίγμα ταφ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε 41 υπέρ 1 εναντίον δεύτερο τμήμα της F σίγμα ταφ άρχεται Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 41 υπέρ, 1 εναντίον. Τροπολογία 251. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε 5 υπέρ 38 εναντίον. 252 τροπολογία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 15 υπέρ, 28 εναντίον. Συμβιβασμός I, θ, 9. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 39 υπέρ, κανένας εναντίον. Συμβιβασμός H, ο συμβιβασμός H είναι ο ΙΤΑ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 40 υπέρ 2 εναντίον. Συμβιβασμός G στη συνέχεια. Ζ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 41 υπέρ 2 εναντίον η άλλη καταπίπτει. Συμβιβασμός J στην συνέχεια, J, άρχεται, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός K, J, α, άρχεται, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 37 υπέρ 2 εναντίον. Συμβιβασμός L στη συνέχεια. ΙΒ άρχεται. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 40 υπέρ κανείς εναντίον. Η επόμενη τροπολογία είναι η τροπολογία 6. Τροπολογία 6 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 38 υπέρ 2 εναντίον. Τροπολογία 62 καταπίπτει, η 7 αποσύρθηκε, η 8 καταπίπτει, η τροπολογία 10 τώρα. Άρχεται. Ψηφίζουμε την 10. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 38 υπέρ 5 εναντίον. Τροπολογία 48. 48 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 2 υπέρ 39 εναντίον. Τροπολογία 47. Άρχεται. Μπορούμε ομού να ψηφίσουμε όλες αυτές μαζί. Όχι, όχι, δεν γίνεται ομού. Η 47 λοιπόν ξεχωριστά. Άρχεται. Τώρα λίγη ψηφοφορία. Λίγη σε λίγο. Ολοκληρώστε. Εντάξει, 28 υπέρ 13 εναντίον εγκρίθηκε. Οι άλλες καταπίπτουν. Περνάμε στην τροπολογία 54. Όχι, οι άλλες κατέπεσαν επειδή ε, εγκρίθηκε η προηγούμενη. Πάμε τώρα, όχι πάνε και αυτές, πάμε στο συμβιβασμό M. Συμβιβασμός M ή ΙΓ. Άρχεται, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν 37 υπέρ 4 εναντίον. Τροπολογία 60 τώρα. 61 λέγεται στην πρόεδρο. Κατέπεσε 60, 61 τώρα. Η τροπολογία 61 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Καταψηφίστηκε 17 υπέρ 25 εναντίον. Τροπολογία 63. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Καταψηφίστηκε 22 εναντίον 17 υπέρ. Συμβιβασμός N, δέλτα άρχεται. Εγκρίθηκε. Λίγη ψηφοφορία εννοώ, λέγει η Πρόεδρος, μάλιστα. Τώρα εγκρίθηκε πλέον. Ναι, το μάντεψα αυτό. Πολλά πράγματα κατέπεσαν, όχι όμως η 64. Τροπολογία 64 λοιπόν τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορριφθήκε 17 υπέρ 24 εναντίον. Επόμενη που θα ψηφίσουμε τροπολογία 70. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 3 υπέρ 40 εναντίον. Της απασχόλησης, Επιτροπής Απασχόλησης, τροπολογία 1. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε 23 υπέρ 19 εναντίον. Τη επιτροπή απασχόληση τροπολογία 2. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορία. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 38 υπέρ 4 εναντίον. Τη επιτροπή απασχόληση η 3 καταπίπτει. τη επιτροπή απασχόληση 4. Τροπολογία 4 άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 22 υπέρ 18 εναντίον της απασχόλησης 5, Επιτροπής Απασχόλησης 5 άρχεται. Τέλος ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία έληξε, εγκρίθηκε 20 υπέρ 18 εναντίον. Μετά κατέπεσαν οι άλλες 72 στη συνέχεια. Άρχεται τροπολογία 72. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 25 υπέρ, 18 εναντίον. Τροπολογία 73. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 25 εναντίον 16 υπέρ. Μπορούμε στη συνέχεια 74 και 76 να ψηφίσουμε από κοινού. 74 και 76 από κοινού. Άρχονται. Ψηφίσατε όλοι. Και οι δύο απορρίφθηκαν. 4 υπέρ 39 εναντίον. Στη συνέχεια τροπολογία 77. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ψηφ... Λίγη ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 3 υπέρ 37 εναντίον. Τροπολογία 78. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε 14 υπέρ, 28 εναντίον, τροπολογία 79. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 31 υπέρ, 3 εναντίον. Της απασχόλησης η τροπολογία 7. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 14 υπέρ, 22 εναντίον. Τροπολογία 80. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 30 υπέρ 10 εναντίον. Τροπολογία 81. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. 2 υπέρ 41 εναντίον. τη απασχόληση 8. Employment 8. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκε 14 υπέρ 24 εναντίον τροπολογία 82 καταπίπτει 83 άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκε 2 υπέρ 41 εναντίον τροπολογία 84 άρχεται ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκε 18 υπέρ 23 εναντίον Τροπολογία 85. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 31 υπέρ, 7 εναντίον. Της Επιτροπής Απασχόλησης η τροπολογία 9. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 15 υπέρ, 26 εναντίον. Η τροπολογία 86. Άρχεται. Οι Διερμηνή. Σα ευχαριστούν, αλλά έληξε ο χρόνος διερμηνία μας. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. voted? Votes closing. Right, votes closed. That's carried 32 to 7. Compromise O. What's not working?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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.